Äh, χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας καθώς και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί διατίθενται έχετε αντιρρήσεις όχι άρα θεωρούνται εγκεκριμένα τα συνοπτικά πρακτικά ο Πρόεδρος έλαβε από το Συμβούλιο μια θέση σε πρώτη ανάγνωση